ψυχούν, αλλά θα αισθάνονται σίγουροι ότι οι βασικές αρχές μας παραμένουν και δεν τίθεται ε, σε κίνδυνο. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ε, κύριος Κυρχόπ, για ένα λεπτό. Ε,